Przewodniczący! Witam Państwa e, obecnych na e, kolejnym posiedzeniu. σας ε, χαιρετίζω καρδιότατα και κυρίως στην τέμη της σημερινής μας συνεδρίασης. Ευρωπαϊκή Ράτζε ε, το πρώτο σημείο της ημερησίας διάταξης είναι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου. Δηλώσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής. Σύμφωνα με τις συνδίκηση της Λισαβόνας θα κάνει καταρχήν μια παρουσίαση ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Herman van Rompuy, θα κάνει μια παρουσίαση και σας καλωσορίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Uh, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχηθώ σε όλους ένα ευτυχισμένο νέο έτος. Σας το εύχομαι προσωπικά για σας κύριε Πρόεδρε, αλλά και για ολόκληρη την Ένωση σε αυτούς τους κρίσιμους καιρούς. το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι πίσω μας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι κάθε φορά δίνω μια πλήρη αναφορά σε σχέση με τα αποτελέσματα λίγες ώρες μετά τη συνεδρίαση. Σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ασχοληθήκαμε την πρώτη μέρα με τα οικονομικά θέματα και τη δεύτερη μέρα με τα εξωτερικά. Καταλήξαμε σε κάποια σημαντικά οικονομικά συμπεράσματα. Πρώτα απ' όλα αποφασίσαμε για την πρόταση μιας την πρόταση δημιουργίας μόνιμου μηχανισμού για την εξασφάλιση της σταθερότητας της Ευρωζώνης. Είχαμε συμφωνήσει καταρχή τον Οκτώβριο ότι χρειάζεται μία τροποποίηση της συνθήκης. Συμβουλεύτηκαν λοιπόν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε σχέση με την ενδεχομένη σύνταξη του κειμένου έχουμε δύο φράσεις που θα προσθεθούν στο 136 της συνθήκης και σας διαβάζω. Τα κράτη-μέλη των οποίων το νόμισμα είναι το ευρώ μπορούν να ιδρύσουν ένα μηχανισμό σταθερότητας που ενεργοποιείται όταν είναι απαραίτητο να προστατευτεί η σταθερότητα της ευρωζώνης στο σύνολό της. Και η απαιτούμενη ενίσχυση κάτω από ένα τέτοιο μηχανισμό θα είναι κάτω από αυστηρούς όρους. Και αυτό είναι σημαντικό για να μπορέσει η Ευρώπη να προστατεύεται από τις κρίσεις και αυτό είναι απαραίτητο όχι μόνο για την ασφάλεια του δικαίου αλλά για την αξιοπιστία στην αγορά. Δεν θα ενισχυθούν έτσι οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, συμφώνησαν τα μέλη ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απλουστευμένη διαδικασία τροποποίησης. Τώρα απαιτείται γνωμοδότηση από το Κοινοβούλιο σας καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Κεντρική Τράπεζα. Θέλω να εξασφαλίσουμε την έγκρισή σας. Σας υπενθυμίζω πόσο σημαντικό είναι να προχωρήσετε το ταχύτερο και το ομαλότερο δυνατόν σε αυτό το θέμα, γιατί η ρευστότητα της αγοράς εξακολουθεί να μας ανησυχεί. Ξέρω ότι εσείς και οι επιτροπές σας που είναι υπεύθυνε παρακολουθούν το θέμα από κοντά και κατά τη ε, διάρκεια των συναντήσεων της ομάδας που προείδρευσα είχαμε συναντήσεις με τις προεδρίες των επιτροπών που είναι πιο αρμόδιες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Μπούζεκ για τη συμβολή του και χαιρόμαστε που μας ενημέρωσε ότι το Ευρωκοινοβούλιο θέλει να προχωρήσει γρήγορα όσον αφορά αυτό το θέμα. Με τη γνώμη σας θα μπορέσουμε να συντάξουμε αυτή την απόφαση οριστικά και να εγκριθεί το Μάρτιο. Στη συνέχεια η τροπολογία θα πρέπει να εγκριθεί από όλα τα κράτη-μέλη και θα θέλαμε να τεθεί σε ισχύ το αργότερο 1η Ιανουαρίου 2013 ώστε ο μόνιμος μηχανισμός να τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του μηχανισμού είναι τα εξή. Τον... Είχαμε ζητήσει από την Κομισιό τον Οκτώβριο να κάνει προπαρασκευαστική εργασία και είχαμε μία δήλωση στις 28 Νοεμβρίου που εγκρίθηκε πλήρως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στο μέλλον λοιπόν ο μηχανισμός σταθερότητας θα συσταθεί βάσει του υφιστάμενου μηχανισμού η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να προσχωρεί απόλυτα στα, στους κανόνες και στις πρακτικές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά περίπτωση. Συνεπώς η ιδιωτική συμμετοχή δεν θα είναι προκαταρτικός όρος για το μέλλον του μηχανισμού σταθερότητας. Επίσης, Είχαμε πολύ καλά ανταλλαγέ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε σχέση πώς, με το πώς να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, της μεσοπρόθεσμες και της βραχυπρόθεσμας όλων των ευρωπαϊκών οικονομιών. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ ήταν επίσης παρόν, γίναν δηλώσεις και αυτή η συζήτηση επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα και την ενότητα μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμών. Όλοι γύρω από το τραπέζι ε, συμφώνησαν με τη βασική ανάλυση. Επιμένω ότι και 27 συμφωνούν, έστω και αν η ανάλυση ασχολείται περισσότερο με τα 17 κράτη με το ευρώ θέλουμε οι οικονομίες μας να γίνουν πιο ανθεκτικές στην κρίση και να έχουμε ε, νέα δομή οικονομική στην Ευρώπη. Εγκρίθηκε λοιπόν μία δήλωση. Τρία, σημεία αφορούν τις εθνικές κυβερνήσεις. Φορολογική υπευθυνότητα, δημοσιονομική υπευθυνότητα, ε, ε, ενίσχυση της ανάπτυξης και εφαρμογή αναγκαίων μέτρων η Ελλάδα και η Ιρλανδία καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Τα άλλα θέματα αφορούσαν την εργασία των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων μαζί. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρώτα απ' όλα ζήτησε από τα άλλα όργανα και βεβαίως από το Ευρωκοινοβούλιο να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία που, στην οποία κατέληξαν τον Οκτώβριο με την Task Force να τεθεί σε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι. Αυτό είναι το κοινό μας καθήκον. Δεύτερον, συμφωνήθηκε να γίνουν νέα stress test στον τραπεζικό τομέα ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρη διαφάνεια μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε αποφασισμένοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είναι έτοιμοι καθώς και τα όργανα να κάνουν ό,τι χρειάζεται για την εξασφάλιση της σταθερότητας της Ευρωζώνης, όπως ελέγχθη. Και πραγματοποιείται εργασία πραγματική για να ε, επισπευστούν αυτά. Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησής μας ασχολήθηκαμε με τη σχέση με τους στρατηγικούς εταίρους. Η Lady Άστον υπέβαλε σχετική έκθεση και ενημέρωσα τους συναδέλφους σχετικά με τα θετικά αποτελέσματα τριών διασκέψεων κορυφής την διάσκεψη κορυφής ε, με τον πρόεδρο Ομπάμα όταν οπου άνοιξαν νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη και την ασφάλεια στην διάσκεψη κορυφής με τον πρόεδρο Μετβέντε και συμφωνήσαμε για την προσχώρηση της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και με τον Πρωθυπουργό Σινγκ ε, ε, προχωρήσαμε σε μια ισορροπημένη συμφωνία εμπορίου που ε, ευχόμαστε να τεθεί σε ισχύ το πρώτο εξάμεινο και είχαμε και κοινή δήλωση για το, τη διεθνή τρομοκρατία. Αυτές οι συναντήσεις δείχνουν ότι για τους εταίρους μας δεν είμαστε μόνο μία οικονομική ένωση αλλά και ένας γεωπολιτικός εταίρος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επίσης έδωσε στο Μαυροβούνιο το καθεστώς υποψηφίου κράτους με την πεποίθηση ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έχουν ευρωπαϊκό προορισμό. Επίσης συμφωνήσαμε και για την ακτή του ελεφαντοστού βάσει των όσων είχαν αποφασίσει οι Υπουργοί Εξωτερικών πριν από μερικές μέρες. Δηλαδή πρέπει να γίνουν σεβαστά τα αποτελέσματα των δημοκρατικών εκλογών. Όπως ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 4 Φεβρουαρίου θα ασχοληθεί βασικά με την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ενέργεια και την ασφάλεια την ενεργειακή κυρίως. Το Μάρτιο θα έχουμε την πρώτη άσκηση του αποκαλούμενου Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Δεν πρέπει να είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά μια ανακατανομή συζητήσεων όσον αφορά την κατάσταση της οικονομίας και της δράσης τις σχετικές. Συνάδελφοι, ξέρουμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τον οικονομικό συντονισμό και τον συγκερασμό μέσα στην Ευρωζώνη. Θα εργαστούμε όσο είναι δυνατόν κατά τρόπο πλαισιωμένο και είμαι πεπισμένος ότι θα βρούμε την απαραίτητη συνένεση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Πρόεδρο ξενόματος της Κομισιόν να πάρει το λόγο. Κύριε σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Έχετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εξότιμα μέλη, το περασμένο έτος η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίσε μία σειρά α, δοκιμασιών και η διάσκεψη κορυφή του Δεκεμβρίου απέδειξε ότι είναι αποφασισμένη να αναλάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να πετύχει στόχου μα. Συμφωνώντα ε, να υπάρχει ο μηχανισμός και να ε, προχωρήσει με τη συνθήκη της Ρισταβάνας ε, ότι απέδειξε ότι υποστηρίζει κάθε μέρος που χρησιμοποιεί τα μέσα αυτά. Η Κομισιόν ε, θα εκδώσει την επίσημη της άποψη για την αλλαγή της συνθήκης πριν από διάσκεψη κορυφής την Ερηνή. Η συμφωνία που επιτεύχθη μας επιτρέπει να επιταχύνουμε τις εργασίες μας και η Κομισιόν θα συνεργαστεί με τους Υπουργούς ε, Οικονομικών για να σκεφτεί τα μέτρα υποστήριξης πριν από την Ιερινή Σύνοδο. Ο μόνος μηχανισμός ήταν αυτός που μπορούσε να έχουν κατά νου τα κράτη-μέλη. Απ' την άλλη μεριά θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνος με τη συνθήκη και θα πρέπει να ενδυναμώσει τους κανόνες σταθερότητας και επιτηρήσεις του προϋπολογισμού. Οι αποφάσεις αυτές βασίζονται σε μια σειρά ευρέα μέτρων που αντιμετωπίζουμε για να αντιμετωπίσουμε και την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της και την ανάγκη ανάπτυξης των θέσεων απασχόληση. Το αναγνωρίζει αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο. Η αρχή κρατών κυβερνήσεω του χώρου του ευρώ διευκρίνησαν απόλυτα ότι είναι έτοιμοι να αναλάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα του, της Ευρωζώνης. Ιδίω και παραθέτω εδώ, καλούνται αποφασιστικές δράσεις για να εξασφαλιστεί η σταθερή υποστήριξη μέσω του Ευρωπαϊκού Μέσου Σταθερότητος πριν να τεθεί σε ισχύ ο μόνιμος μηχανισμός. Αυτά ήταν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Επίσης το Συμβούλιο ζήτησε επιτυχημένη έγκριση μέχρι τον Ιούνιο των προτάσεων της ε, Κομισιόν του περασμένου Σεπτεμβρίου για την καλή διακυβέρνηση και τις προτάσεις ε, του, για το 2020 για την επαναφορά στην αηφόρο ανάπτυξη. Την περασμένη εβδομάδα η Κομισιόν συνένωσε όλες αυτές τις διάφορες προτάσεις για να βρεθεί ο τρόπος διαχείρισης και συντονισμού των αλληλεσυνδόμενων συνοικονομικών μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό το θέμα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διακυβέρνησης, όπου εδώ αποδεικνύεται η εργασία της και η διακυβέρνηση αυτή θα πρέπει να δώσει πλήρη απάντηση στην κρίση. Η Κομισιόν το είπε αυτό ξεκάθαρα στην ετήσια ε, έκθεση για την ανάπτυξη. Γιατί τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξετάσουμε τα επόμενα βήματα. Η πολιτική της οικονομική διακυβέρνηση και συντονισμού έχει αλλάξει. Και όχι μόνο επειδή κάποιοι ομοσπονδιακοί όπως λέγονται το ήθελαν, οι αγορές το ήθελαν, οι διεθνή μας εταιροί το ήθελαν. Είναι θέμα κοινού νου. Και εμείς θα ακολουθήσουμε. Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συνδέουν αυστηρά φορολογικά μέτρα και οικονομικό συντονισμό. Προσφέρουν εκ των προτέρων συντονισμό, συζητώνε δηλαδή η απόψη των μεν και των δε και οικονομικά και ε, φορολογικά πριν προφορήσουμε σε κάποιες ε, βελτιώσεις. Αυτό είναι ένα ιστορικό βήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά χρησιμοποιούμε μια γενική ευρωπαϊκή διάθεση στην οικονομική μας πολιτική. Από εδώ και μπρος θα είναι καλό να ορίζουμε τις πολιτικές από τον προτέρων, όχι να τις ελέγχουμε και να τις συνορίζουμε από τον υστέρων. Βέβαια, γι' αυτό χρειάζεται η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι σωστό αυτό. Η νέα αυτή μορφή της οικονομικής διακυβέρνησης αντικατοπίζει τη νέα πραγματικότητα όταν βλέπουμε το επίπεδο αλληλένδεσης στον ευρωχώρο, στον ναι. Και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προθέσεις που υπάρχουν. Να υπάρχει έτσι με την αλλαγή απόψεων η ενίσχυση των κυβερνήσεων. Λοιπόν, η ετήσια μας έκθεση για την ανάπτυξη προωθεί τις απόψεις αυτή να επανέλθει η σταθερότητα, να επιταχυνθούν τα μέτρα για την ενδυνάμωση της ανάπτυξης. Εάν δεν έχουμε ισολογισμό και ισορροπία, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε νέα ανάπτυξη τη εμπιστοσύνη. Και αν δεν έχουμε εμπιστοσύνη, θα υπάρχει αστάθεια και ε, κοινωνικές επιπτώσεις, Ιδίω όσον αφορά την απασχόληση. Βέβαια, παγίωση φορολογική δεν σημαίνει μόνο η μείωση του χρέους. Σε πολλές ε, τομείς, καινοτομία, παιδεία, νέες μορφές ενέργειας είναι υποψήφιοι για αυτές τις προτεραιότητες. Οι άλλες φασικές ιδέες είναι οι θεσ, ε, θεσμικές ε, αλλαγές. Εμείς θέλουμε να αποφασίσουμε αν θέλουμε ανάπτυξη χωρίς απασχόληση ή ανάπτυξη της απασχόλησης. Εάν είναι το δεύτερο θα πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε μεταρρυθμίσεις της αγοράς απασχόλησης. Θα πρέπει να φροντίσουμε να εργαστούν, να βρουν εργασία εκεί οι άνεργοι με το να κάνουμε την εργασία πιο ελκυστική. Και θα ήθελα να είμαι σαφής εδώ. Η διαρθρωτική μεταρρύθμιση δεν σημαίνει ότι θα μειωθεί το επίπεδο κοινωνικής προστασίας αλλά σημαίνει να μπορέσουμε να εντάξουμε εκείνους που αυτή τη στιγμή αποκλείονται από την αγορά εργασίας, ιδίως τους νέους. Τα επίπεδα ανεργίας σε ορισμένα κράτη-μέλη και σε καλούς καιρούς είναι σκανδαλώδη. Δεν μπορεί και να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, με αυξανόμενο οικονομικό διεθνή ανταγωνισμό, θα πρέπει εμείς να προσαρμόσουμε και την αγορά εργασίας μας. Το πρόγραμμα Ευρώπη 2020 είναι πάρα πολύ κεντρικό για αυτές τις προσπάθειες για να υπάρχουν οικονομικά ωφέλη μέσω και βρέχει πρόθεσμα. Αυτό σημαίνει επένδυση σε τομείς ανάπτυξης και ανάπτυξη ε, του δυναμικού που έχουμε, επενδύσεις στην ενέργεια, στις μεταφορές, στις καινοτομίες. και να προχωρήσουμε προχωρήσουμε στην πίωση για το γύρο της Ντόχα προωθώντας ε, εμπορικές ε, συμφωνίες με τους εταίρους μας. Το, ε, ο επόμενο προλογικό τη Ένωση θα πρέπει να είναι ένα προπολογισμό που θα ενισχύει την ανάπτυξη. Κυρίε και κύριοι, η οικονομία τώρα κινείται προ την σωστή κατεύθυνση. Φέτος, θα πρέπει να υπάρχει αύξηση του ΟΕΠ της τάξης του 1,5% και 2% το 2012. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει βελτίωση της απασχόλησης. Χάρη ιδίω στα μέτρα παγίωσης που υιοθετήθηκαν, υιοθετήθηκαν ήδη. Το έλλειμμα προβλέπεται να μειωθεί από το 6,8% στο 4,2% το 2012. Για να μπορέσουμε όμως να ανακουφιστούμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει αλλάξει ο κόσμος. Δεν μπορούμε να περάσουμε στις παλιές μεθόδους. Εν ώψη της ε, μεγαλύτερης κρίσης ε, του Ευρωπαϊκής Ένωσης από τότε που ιδρύθηκε θα πρέπει να υιοθετηθούν επιτέλους τα σωστά μέτρα. Εάν δεν υιοθετηθούν αυτές οι αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να το κάνουμε εμείς. Δηλαδή, μόνο με την επίλυση του χρέους και σταθεροποίηση των οικονομικών θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ανάπτυξη. Και όχι τυχαία ανάπτυξη, αηφόρο ανάπτυξη, που θα περιλαμβάνει όλους. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, υπάρξουν μεταρρυθμίσεις που προωθούμε εδώ και πολλία χρόνια. Μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν τις τιμές και θα βελτιώσουν τις ευκαιρίες για νέους τρόπους αντιμετώπισης της ενεργείας. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να το κάνουμε. Η ετήσια έκθεση ανάπτυξης κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε σε μια οικονομική ε, έναν οικονομικό συνολισμό και πραγματική διακυβέρνηση οικονομική για όλους τους ε, πολίτες. Ευχαριστώ. On of the... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος του ΕΛΚ, ο Πρόεδρος κ. Ντόλν. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Κομισιόν, το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το κατέδειξε. Το το ευρώ είναι ένας πυλώνας σημαντικός για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση και όλα θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να σταθεροποιηθεί και να ενισχυθεί. Οι αργοί κρατών και κυβερνήσεων επιβεβαίωσαν την δέσμευσή τους στο ευρωπαϊκό νόμισμα και την προσχώρηση της Εστονίας στις αρχές του έτους αποτελεί ένα επιπλέον δείγμα προς την κατεύθυνση αυτή και θα έλεγα ένα πολύ καλό μήνυμα για το πώς μπορούν να τηρηθούν τα κριτήρια για τις μεγάλες χώρες που δεν τα τηρούν. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε όμως ότι όλοι γνωρίζουμε την τεράστια οικονομική κρίση που διανύει η Ευρώπη στο, και ιδιαίτερα οι χώρες ευρώ. Θα πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια το 2010 για να ξεπράξουμε προβλήματα, να, να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία μας και να καθυσυχάσουμε τις αζαγίες, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για απασχόληση και ανάπτυξη μακροπροθέσμους. Νομίζω ότι εδώ μιλάμε την ίδια γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι τα δημοσιονομικά σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να εξηγιανθούν και να μην ε, πάψουν οι προσπάθειες. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συγκλίνουν και να συντονίσουν τις δημοσιονομικές πολιτικές αλλά και τις νομισματικές πολιτικές. Αυτό σημαίνει πως χρειάζεται να συμφωνήσουμε για τα ταμεία ενίσχυσης της ζώνης ευρώ και αυτό έχει σημασία και έννοια μόνο εάν εφαρμοστούν οι κανόνες. Οι πολίτες μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να ε, γίνει πολύ ασφαιρή διαχείριση των δημοσιονομικών, διαφορετικά δεν ε, θα μπορέσουν να ξεφύγουν από τον τεφαύλο κύκλο. Να ε, δημιουργήσουμε προποθέσει για ανάπτυξη και απασχόληση. Το αναφέρατε και εσείς, να ολοκληρώσουμε την ιστορική αγορά, να επενδύσουμε περισσότερο στην, στην έρευνα και την κατάρτιση και την διαβίου κατάρτιση. Η ομάδα μου επιθυμεί η κινητική προσέγγιση να ευνοηθεί στο σχέση με την προσέγγιση την ε, διακυβερνητική, διότι θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικέ τράσει μα. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, σα ζητώ να διασφαλίσετε πω η μεταρρύθμιση τη συνθήκη που βιώθηκε στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Και έπειτα μια δημοσιονομική συζήτηση, η οποία μόλι ξεκινάει, να πω ότι η ομάδα μου θα συνεχίσει να μιλάει για μια διευθέτηση των δημοσιονομικών στο αγγείς μέλλον προκειμένου να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις απασχόλησης και ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αγαπητέ Πρόεδρε της Κομισιόν, θα πρέπει να μην φοβηθούμε, να λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα και να πάρουμε ένα, δύο, τρία παραδείγματα στον προπολογισμό 1%, 2%, 5% τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να εξέλθουμε αυτή την κρίση. Δεν μπορούμε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα εάν δεν έχουμε περισσότερα κονδύλια. Αυτό σημαίνει ότι τα κρατημέλη χρειάζεται να δαπανίσουν περισσότερα χρόνια. Μην φοβούστε, Πρόεδρε Βανδρόμπο και κύριε Μπαρόζο. Κάντε μας ε, αυτές τις προτάσεις και αργή κρατών κυβερνήσεων από κοινού, με το Κοινοβούλιο θα φροντίσουν να βρουν την κατάλληλη λύση, τη σωστή λύση, αλλά τουλάχιστον έχουμε μπροστά μα ε, πολλέ. Ε, πολλά παραδείγματα και δυνατότητες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Στίβεν Χιούς έχει το λόγο εξ ονόματος των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου μας έδωσε μια πολιτική συμφωνία σχετικά με τον μηχανισμό επίλυσης της κρίσης. Οι αντιδράσεις των αγορών μετά τις αγορές ε, δείξαν ότι υπήρχαν διάφοροι φόβοι για την Πορτογαλία, την Ισπανία και το Βέλγιο. Θα πρέπει να ρωτήσουμε για ακόμα φορά αν αυτά τα οποία έγιναν, έγιναν αργά και ε, δεν έγιναν σε βάθος. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρξει σταθεροποίηση των ε, χρήματα και ο νέος ε, μηχανισμός θεωρείται τώρα ως ανεπαρκής. Χάσαμε λοιπόν μια ακόμα ευκαιρία και το Δεκέμβριο το Κοινοβούλιο έστειλε ένα σήμα για το ευρωομόλογο από το Συμβούλιο αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση ούτε από το Συμβούλιο ούτε από την Κομισιόν. Από το 2008 συνεχίζουμε να επαναλαμβάνουμε αυτά τα θέματα και να τονίζουμε τη σημασία που έχουν και κάθε φορά η απάντηση που λαμβάνουμε είναι πολύ μικρή και σίγουρα πολύ χαμηλότερη των περιστάσεων. Στον... Στις νομισματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεν έχουμε τις, τα απαραίτητα ε, μέσα και εργαλεία για να τις αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει ταυτόχρονα έλλειψη μιας ε, σωστής δημοσιονομικής πολιτικής. Οι ε, αγορές δεν ασκούν μόνο πίεση λόγω του υψηλού χρέους και των υψηλών ελλημάτων, κύριε Μπαρόζο. Το πράττουν διότι επιθυμούν να έχουν διασφάλιση των χρημάτων τα οποία δανείζουν. Τι κρατάει την ε, Ευρωζώνη σήμερα ενωμένη. Είναι το, ο φόβος της κατάρρευσης του συστήματος. Νομίζω ότι δεν μπορέσε να ανταποκριθείτε στην κρίση και αυτό οδηγεί στην, την Ευρώπη σε, μια, σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Αυτό που είναι απαραίτητο τώρα είναι να υπάρξουν ε, οι κατάλληλοι θεσμοί μέσω της αναθεωρημένης ε, συνθήκης ο επικεφαλής της ε, Bundesbank, Bundesbank δεν ε, επιθυμεί ενδεχομένω να συμβεί κάτι τέτοιο και να πω επίσης κύριε Μπαρόζο ότι υπήρξαν επιθέσεις ε, από το εξωτερικό όπως γνωρίζετε ιδιαίτερα κατευθυνόμενες κατά της Ιρλανδίας χρειάζεται λοιπόν να εργαστούμε για να προστατεύσουμε και τις θέσεις απασχόλησης αλλά και τα δικαιώματα των εργαζομένων και να συνεχίσουν να ισχύουν οι συλλογικέ συμβάσει. Εάν δεν το πράξουμε αυτό, σίγουρα θα επηρεάσουμε αρνητικά το ευρωπαϊκό όραμα. Ε, οι λαοί μας δεν θα δεχθούν μια αποτυχία. Ο κ. Φάρατζ ε, νέφει καταφατικά. Ο πρόεδρος ε, Μπαρόζο νομίζω ότι δίνει ε, κάποια βέλη στην ε, φαρέτα του κυρίου Φαρέτα. Ευχαριστώ συνάδελφε. Η κυρία Σιλβίγκουλα εκ μέρους των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τα συμπεράσματα του, Δεκεμβρίου, του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Πρώτο σχόλιο. Η κρίση έχει ιδιαίτερη επίδραση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μια κοινότητα δικαίου εξ αρχής και επειδή είμαστε μια κοινότητα δικαίου, ο κανόνας είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Συνεπώς θα τηρήσουμε τον κανόνα. Αλλά όταν αντιμετωπίζουμε μια κρίση τόσο βαριά όπως το υπενθυμίζει ο πρόεδρος το Annual Growth Survey το παρατήρησε πρέπει να ενεργήσουμε και όχι να νομολογούμε. Λέτε ότι η ε, τροποποίηση της συνθήκης είναι απαραίτητη για να ε, ηρεμήσουν οι αγορές. Πρώτα απ' όλα, με συγχωρείτε, αλλά μετά το το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου δεν αισθάνθηκα οι αγορές να εφησυχάζουν. Λοιπόν, προσέξτε πώ θα τι κάνετε να ησυχάσουν. Αλλά για φανταστείτε τι θα συμβεί αν αποτύχει η τροποποίηση. Είχαμε στη χώρα μου ένα αρνητικό δημοψήφισμα και ήσασταν ήδη εκεί κύριε Μπαρόζο. Καμιά φορά πρέπει να σκέφτεστε όταν λέμε στην αγορά ότι πρέπει να τροποποιήσουμε τη συνθήκη. Όλα πρέπει να γίνουν μέχρι τάδε ημερομηνία και ελπίζουμε. Βεβαίω ε, επιλέγετε την απλουστευμένη διαδικασία ελπίζοντα ότι θα περάσει. Αλλά αν περάσει θα ησυχάσουν ίσως οι αγορές αλλά σίγουρα όχι οι λαοί. Έρχομαι στο δεύτερο σχόλιο. Πολύ φασαρία για το τίποτα αλλάζετε τη συνθήκη για ένα θέμα δικαίου. Δεν τη μεταβάλλετε τη συνθήκη για να δώσετε στους πολίτες τις απαντήσεις που περιμένουν. Και εμεί είμαστε οι εδώ. Εξετάζουμε την κυβερνητική διακυβέρνηση και συμφωνήσαμε ε, να έχουμε σταθερή συνθήκη. Αλλά τώρα στο δρόμο μας λέτε ότι θα τροποποιήσουμε τη συνθήκη. Τι θα γίνει λοιπόν. Θα πούμε στους πολίτες ότι θα τροποποιήσουμε τη συνθήκη. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα δικαίου, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να τους δώσουμε δουλειά. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου μας ζητά να επισπεύσουμε. Ωραία, ας επισπεύσουμε, λέει κύριε Βαν Ρόμποϊ, ε, α επισπεύσει και το Συμβούλιο. Υπάρχει απλό τρόπο να γίνει αυτό. Να προσεγγίσετε στι θέσει μα και να σταματήσετε να θεωρείτε τη συναπόφαση ε, σαν ε, να πρέπει πάντα το Ευρωκοινοβούλιο να προσαρμόζεται. Τη διακόπτη την κυρία ο Πρόεδρος. Η κύριε Συμπρόεδρος των Πρασίνων, η Ρεμπέκα το Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αυτό που εγώ θυμάμαι από την τελευταία διάσκεψη ε, κορυφής δεν παρουσιάστηκε στην δική σας ε, παρουσίαση. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των Βρυξελών η εταιρεία εξολόγησης Moody's μείωσε την ε, ταξινόμηση για την Ιρλανδία. Αυτό ήταν ε, μία απόδειξη πόσο μεγάλη είναι η αποτυχία μας μέχρι στιγμής σε σχέση με την κρίση που μας απασχολεί σήμερα και που μας απασχολεί μέσα στην σύγκριση αυτή τη διεθνή των στοιχείων ε, είναι να απορεί κανένας πώς ε, επιτυχής είναι η κερδοσκοπία αυτή τη στιγμή έναντι του ευρώ ενώ μια χώρα που έχει μεγαλύτερα προβλήματα από την Ισπανία, από την Πορτογαλία ή είπα δηλαδή δεν ε, πλήττεται από τις επιθέσεις αυτές των κερδοσκόπων. Αυτή είναι η δηλαδη δεν πληττεται Ξεκινήσαμε ένα καινούριο έτος έχουμε καινούργια προβλήματα επιτάπητος. Αυτό που είπαμε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ότι δεν επαρκεί αυτό που αποφασίστηκε θα πρέπει να είναι αυτό που θα με απασχολήσει εδώ και τώρα. Πιστεύω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται με τα τεράστια χρέη και ιδιωτικά χρέη αλλά και απαράδεκτο δημόσιο χρέος πολλών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που από μόνο τους δεν θα μπορέσουν να βγουν από την κρίση. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Θεωρούμε ότι η μείωση του δημοσίου χρέους όπως έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή σε διάφορα κράτη-μέλη όπως έχει ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Συμφωνία των κρατών μελών δεν αρκεί και τα κράτη-μέλη φτάνουν στα όρια του αποδεκτού. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια νέα συνεννόηση πώς θα μπορέσει να θεωρηθεί αυτό επαρκές. Η εξέλιξη στην Ουγγαρία είναι πραγματικά ανησυχητική. Όταν βλέπουμε τις ε, διαφορές που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών γιατί όταν μειώνεται το δημόσιο χρέος θα πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου, να είμαστε πιο δίκαιοι και λέω ρητά ότι ο τραπεζικός τομέας πρέπει να αναδιαρθρωθεί δεν είμαστε πεπισμένοι ότι με την διάσωση τον ε, του χρέους ε, αυτή τη στιγμή που μετατοπίζεται απλώς θα μπορέσει να βρεθεί μια πραγματική λύση. Και χρειαζόμαστε μια προοπτική μέσα στα πλαίσια ενός νέου πράσι, μιας νέας πράσινης συμφωνίας και να μπορέσουμε έτσι να ξεκινήσουμε μια νέα ε, άγουσα. Είναι θαυμάσια πατρίδα η Ευρώπη, θα το τονίσω αλλά πριν πολύ να κάνουμε να το διατηρήσουμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Συντηρητική και ο κύριος Κυρκόπ έχει το λόγο. Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε σημαντικέ αποφάσει για τη μελλοντική διαχείριση κρίσεων. Αλλά συμφωνώ με τον Πρόεδρο Παρόσο ότι παραμένουν τα προβλήματα. Πρέπει να επανέλθουμε σε δημοσιονομική πειθαρχία και ορισμένε χώρε δεν προχωρούν σε οικονομική μεταρρύθμιση. Μου είπαν, ότι με ένα ενιαίο νόμισμα δεν μπορεί κανεί να υποτιμήσει για να βγει από την κρίση. Πρέπει να μεταρρυθμίσει την οικονομία του για να προχωρήσει Πολλοί από εμά είχαν δίκιο που δεν μπήκαν στο ευρώ. Ορισμένα κράτη-μέλη μπόρεσαν να βρουν άλλε λύσει για να ενισχύσουν τεχνητά ε, την οικονομία τους ε, αποτιμώντα υπερβολικά ψηλά το ενεργητικό τους και μην παίρνοντα διορθωτικά μέτρα ή βάζοντας δημόσια χρήματα σε περιπτώσεις που δεν αποδίδουν και μάλιστα οδηγούν σε ε, δημοσιονομικό έλλειμμα. Βεβαίω πρέπει να βρούμε λύσει για να αντιμετωπίσουμε τις άμεσες επιπτώσεις αυτής της πολιτικής ε, φορολογική σταθερότητα είναι σημαντική, πρέπει όμως να δημιουργήσουμε ευκαμψία στην αγορά εργασίας, να ανοίξουμε τις αγορές, να καταργήσουμε τα εμπόδια στο εμπόριο, να υποκινήσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία, ώστε ε, να μπορέσουμε να μειώσουμε τις δημόσιες δαπάνες υπήρξε μεγάλη παρέμβαση ε, του δημοσίου στην οικονομία, αλλά αυτό είναι ανακουφιστικό, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Χρειαζόμαστε οικονομική ανάπτυξη και επιτυχημένες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες μέσα σε ανταγωνιστικές αγορές, ώστε να, να αποδοθεί αξία στον καταναλωτή και να ισορροπήσουμε. Η ε, Single Market Act και καινοτομία είναι πολύ σημαντικές και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε την απαραίτητη προσοχή. Ε, άλλες χώρες τώρα στον κόσμο με διαφορετικές αξίες έχουν προχωρήσει. Εάν δεν βγούμε προοδευτικά από αυτή την κρίση θα βρεθούμε σε παρακμή και θα είναι πολύ σημαντικές οι επιπτώσεις όσον αφορά την προώθηση των αξιών μας και θα επηρεάσουμε και το μέλλον του πλανήτη. Ευχαριστώ για την ομιλία σας. Ο κύριος Τζο Higgins, Ενωμένη Αριστερά. Στην πρακτική ο μηχανισμός σταθερότητας δεν είναι παρά ένα άλλο εργαλείο για να προστατευτούν οι τράπεζες της Ευρώπης από την φοβερή τους κερδοσκοπία. Είναι ένας μηχανισμός ε, που καθιστά την εργαζόμενη τάξη της Ευρώπης υπόχρεη να πληρώσει την κρίση του καπιταλισμού. Ε, ε, κύριε Μπαρόσο και Βαν Ρόμπαϊ, ε, μας λέτε σήμερα σας παρακαλώ ποια είναι η δοντολογία της μεταφοράς εκατομμυρίων ευρώ χρεών του ιδιωτικού τομέα στους ώμους, μεταφορά αυτών των χρεών στους ώμους του Ιρλανδικού λαού που δεν έφταιγε σε τίποτα η παρέμβαση του Δούνου του και της Ευρώπης στην Ιρλανδία ουσιαστικά καθιστούν τους Ιρλανδούς φορολογούμενους δούλους. Καταστρέφεται τις υπηρεσίες και το επίπεδο διαβίωσης των λαών. Λέτε ότι είσαστε δημοκράτες, αλλά υποδουλώνετε τους Ευρωπαίους στις χρηματοπιστωτικές αγορές που σας που σας σέρνουν από τη μύτη. Ο μηχανισμός σας είναι ένα άθλιο εργαλείο το οποίο σας το υπαγορεύει η αγορά και θα επιμείνουμε να πάμε σε δημοψήφισμα στην Ιρλανδία προτού περάσει οτιδήποτε. Ο κύριος Νάιτζελ Φάρατζου. Ευχαριστώ. Τι όρο χρησιμοποιούμε συνήθως στη σύνδεση με την, ε, με την Ευρώπη. Δεν είναι αποτυχία, αλλά σταθερότητα δεν καθελέγαμε ότι όταν θα έχουμε το ευρώ θα έχουμε και σταθερότητα. Θα πρότεινα λοιπόν από εδώ και στο εξή ε, να μιλάμε για χάος και για αθλειότητα. Ο όρος σταθερότητα όμως συνεχίζεται να χρησιμοποιείται σήμερα και από τον κύριο Βανδροπόη και από τον κύριο Μπαρόζο. Σταθερότητα <clears throat> όμως δεν υπάρχει. Το βλέπουμε στην Πορτογαλία και την περσμένη εβδομάδα. Ήταν Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα με χρήματα των φορολογουμένων εξαγόραζε χρέος. Βλέπετε λοιπόν ότι το σύστημα δεν λειτουργεί. Νομίζω λοιπόν ότι αστείευεστε κύριε Ρομπόη. Χθε ε, τα επιτόκια ανέβηκαν σημαντικά στην ε, Πορτογαλία και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η μάχη για την Ισπανία. Αυτό το οποίο θέλετε να κάνετε είναι να διπλασιάσετε τα κονδύλια που πρόκειται να χορηγηθούν στην διάσωση των τραπεζών. Χρησιμοποιείται λοιπόν την κρίση ως έναν τρόπο για να μας καθοδηγήσει τη συγκεκριμένη μουσονομική πολιτική στην Ευρώπη. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε σήμερα είναι να μην μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά για Ένωση υπερχρεωμένη. Χρειάζεται λοιπόν η πολιτική σας είναι αυτή που οδηγεί στην φυλάκιση των ε, χωρών του Νότου και θα αναγκαστείτε να πληρώνετε αιωνίως ε, για την διάσωση αυτών των οικονομιών. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο όπου δεν έχει καμία σημασία αυτά τα οποία λέτε. Κανείς δεν σας πιστεύει, το κοινό δεν σας στηρίζει και οι αγορές συνεχίζουν ε, να κρυμνίζονται. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαντλένερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, ωραία λόγια, αλλά κενά περιεχομένου από τον κύριο Μπαρόζο. Άκουσα ότι οι πλούσιοι πληρώνουν για τους ε, αδύναμους. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα συνεχιστεί εδώ και για πολλά χρόνια. Πρέπει να διασώσουμε τις χώρες αυτές. αλλά το πώς θα γίνει αυτό δεν ε, μας λένε. Παίρνουμε χρήματα από τους Ολλανδούς πολίτες οι οποίοι πρέπει να πληρώσουν τις άλλες αδύναμες χώρες που εισήλθαν στο ευρώ δολίως θα, τι θα πρέπει να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε δεν ακούμε τίποτα γιατί να μην ε, έχουμε ένα σενάριο ώστε χώρες όπως η Ελλάδα να επιστρέψουν στην ε, εθνικό του νόμισμα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να προβλέψουμε ένα τέτοιο σενάριο. Αυτό το λένε όλοι οι οικονομολόγοι. Είναι η καλύτερη λύση κατά την άποψή του. Τώρα, για την ε, απασχόληση. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να την στηρίξουμε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει. Ε, ζητάει από την Ολλανδία περισσότερη σύνδρομη συνεισφορά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Λοιπόν, με λίγα λόγια θέλω να πω ότι κάτω χώρε πληρώνουν για τις αδύναμες και για τις χώρες με αδύναμες οικονομίες υπάρχουν 27 δισεκατομμύρια τα οποία έχουμε καταβάλει για το Ταμείο Διάσωσης ε, των ε, Αδυνάμων Χωρών. Οι δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνονται, ενώ εμείς ε, χρειάζεται να εξοικονομήσουμε και να εξηγιάνουμε τις οικονομίες μας. Αυτή η οικονομική Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, είναι, δεν γίνεται μάλλον Άρχισα να παρατηρήσω ότι υπήρχε μια και μπλε κάρτα για τον κύριο Φάραντ. Θέλετε να βάλετε μια ερώτηση. Συνήθως χρησιμοποιώ τη μετρική μου γλώσσα, αλλά καμιά φορά είναι διασκεδαστικό να ακούει κανένας τον κύριο Φαράζ, γιατί ξέχει όλες τις απαντήσεις τις ερωτήσεις που ο ίδιος ε, δίνει. Αλλά ποια είναι η εναλλακτική, κύριε Φαράτζο. Αν είχαμε 16 έως 20 διαφορετικά νομίσματα όπως είχαμε την δεκαετία του 90 όταν κατέρευσε η Βρετανική Λύρα θα ήταν καλύτερο. Αυτό θα είχε βελτιωθεί η κατάσταση στην Ευρώπη. Κανένας οικονομικός, κύριε Φαράτζ θα μπορούσε να συμφωνήσει με αυτό. Δεν μπορείτε να πείτε ότι ζούμε στο παρελθόν. Όχι, αντιμετωπίζουμε θέματα που αφορούν την Ευρώπη τη σήμερα και εσείς ποτέ, ποτέ κύριε Φαράτς, δεν ε, τίθεται το θέμα πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη σημερινή κατάσταση και το μέλλον. Είναι πολύ εύκολο αυτό που κάνετε. Did say a decade ago. Πριν από μια δεκαετία δεν είπα ότι μπορείτε να ενώσετε την Ελλάδα και τη Γερμανία στην ίδια νομισματική ένωση και θα λειτουργούσε αυτό. Και αν εξετάσετε την ιστορία θα δείτε ότι αν ενώνονται άτομοι υποχρεωτικά σε ενώσει, όταν οι κυβέρνηση νομίζουν ότι ξέρουν τα πράγματα καλύτερα από τι αγορέ, πάντα χάνουν οι κυβερνήσει. Με ρωτάτε ποια είναι η λύση μου σήμερα είναι απόλυτα σαφής. Η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ελλάδα δεν ταιριάζουν μέσα στην Ευρωζώνη. Και αυτό θα πρέπει να κάνουμε, αυτό θα πρέπει να κάνει ο κύριος Φον Ρόμποϊ, είναι να εισάγει ένα πρόγραμμα για να επιτρέψει στις χώρες αυτές να επανέλθουν στο δικό τους ε, νόμισμα, να έχουν ε, υποτίμηση ανταγωνιστική και να έχουν αθέστα απασχόληση. Γιατί αυτή η πολιτική σκοτώνει τις αγορές. Ο κύριος Μαρσία Μαργκάγιο, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αν διαβάσετε τα περιοδικά σήμερα θα κάνετε δύο διαπιστώσεις. Βρισκόμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο του εθνικού χρέους και ε, προτείνονται μια σειρά από μεμονωμένες δράσεις. Μόνο αυτή τη στιγμή έχουμε ε, το ευρωπαϊκό εξάμεινο, το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης, ε, το σύστημα της ε, διάσωσης, τα ευρωομόλογα για την κάλυψη του εθνικού χρέους, αλλά με, έχουμε επίσης και τα ε, προγράμματα τα συγκεκριμένα και την έκδοση ενδεχομένων ομολόγων για τη χρηματοδότησή τους. Όλα αυτά λοιπόν μπορούμε να τα συνδυάσουμε, θα πρέπει να υπάρξει ένα τελικό σχέδιο για να το παρουσιάσουμε και στους πολίτες. Αυτό το σχέδιο λοιπόν θα πρέπει να είναι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο, ένα σχέδιο το οποίο δεν θα χωρίσει την Ευρώπη στα δύο και στις ε, Ευρώπη των δύο ταχυτήτων, ένα σχέδιο το οποίο θα φροντίσει να πετύχει τους στόχους των ε, δημοσιονομική σταθερότητα και την ε, οικονομική ανάπτυξη για να ξεπεράσουμε την κρίση που αντιμετωπίζουμε. Τώρα, κάτι σχετικά με τον μηχανισμό διάσωση που αναφέρεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. Υπήρξε μια πρώτη δήλωση η οποία έλεγε ότι ε, γινόταν συμμετοχή των ιδιωτών στο ταμείο αυτό, κάτι το οποίο αντίθετο τον πρόεδρο του Κεντρικής Τράπεζας ε, ε, θα πρέπει λοιπόν, όπω είπατε, να εξεταστεί κατά περίπτωση. Ποιο θα αποφασίζει, με τι κριτήρια όμω, τη συμμετοχή ιδιωτών, θα ακολουθούν τα κριτήρια της, ε, του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Η μόνη περίπτωση στην οποία το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο έκανε μια τέτοια παρέμβαση ήταν στην Αργεντινή 2003 και οδήγησε την χώρα σε ένα χάσο το οποίο δεν έχει ακόμα εξέλθει και δεν έχουν ακόμα πληρωθεί ή διοξευληθεί οι ιδιώτες. Θα ήθελα να πω ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια αγορά όπως αυτή των Πολιτειών. θα δώσει μια μεγαλύτερη ρευστότητα, θα μπορέσουν οι τράπεζες να ε, χειριστούν την ρευστότητα αυτή με τις επενδύσεις, αλλά παράλληλα διακόπτει ο πρόεδρος κυρία Μπέρες έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, δεχθήκατε να προεδρεύσετε μια ομάδα λεγόμενη σοφών. Συμμετείχαν υπουργοί οικονομικών που απειλούνται από την επιδίνωση του εθνικού τους χρέους θα μπορούσε να, όλοι αυτοί να αποτελέσουν ε, μια ομάδα σοφών η παραφωνία που υπάρχει ανάμεσα στον πρόεδρο Τρισέ, τον πρόεδρο Μπαρόζο, την κυρία Μέρκελ και τι αγορέ μα λένε ότι δεν προκείτο για μια ομάδα σοφών. Κληθήκατε να διαχειριστεί την κρίση του ευρώ. Έχουμε ανάγκη να διαχειριστούμε το ευρώ προ όφελο των πολιτών τη Ευρώπη και όχι προ όφελο των κερδοσκόπων. Γι' αυτό δεχτήκατε μια μεταρρύθμιση βολική της ε, συνθήκης ε, ενώ ε, είχε υποθεί ότι μια τέτοια μεταρρύθμιση δεν είναι απαραίτητη, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος του Eurogroup. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, μας ε, καλείται να ακολουθήσουμε έναν δρόμο που θα μας οδηγήσει στον δρόμο του πολύ λίγο, πολύ αργά, διότι θα φτάσει η στιγμή όπου θα έχετε την ανάγκη τη σοφία αυτού του Κοινοβουλίου <coughs> προκειμένου να αναθεωρηθεί η συνθήκη, έτσι αύριο να έχουμε μια ε, ε, δημοσιονομική εναρμόνιση, μια φορολογική εναρμόνιση, δάνεια για να διαχειριστούμε με κοινό τρόπο τα χρέη για να συντονίσουμε τι οικονομικέ πολιτικέ. Και αν θέλετε μεταρρύθμιση των συνθηκών, τότε παχιάστε τον τάβρο από τα χέρατα και εφαρμόστε μια ενισχυμένη συνεργασία για τη ζώνη ευρώ για να διαχειρίσετε τα προβλήματα και τι ευθύνε των κρατών αυτή τη ζώνη και να μην αφήσετε να, να διακυμαίνονται και να επηρεάζονται από τι χρηματαγορέ. ευχαριστώ, κυρία μου. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ήταν πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της, αν και ευτυχώ η χώρα μου δεν συμμετέχει στην Ευρωζώνη, τουλάχιστον ε, καλωσορίζω κάποια από τα μέτρα που συμφωνήθηκαν στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα κράτη της Ευρωζώνης πρέπει να είναι υπεύθυνα για να λύσουν τα προβλήματά τους. Χαίρομαι επίσης και για την αναγνώριση, καθυστερημένη βέβαια, του, ε, εκ μέρου του Συμβουλίου ότι το άρθρο 122 είναι τελείως ακατάλληλο για την διάσωση. Ε, δεν πρόκειται για φυσικές καταστροφές βεβαίως. Ετοιμάζοντας λοιπόν αυτό το νέο μηχανισμό ε, που θα τεθεί σε ισχύ το 2013 δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε μια κρίση τώρα. Η κατάσταση είναι πολύ ανησυχη... Ε, ε, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, ενδεχομένω και στο Βέλγιο. Όσον αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι η επιρροή, η επίδραση μάλλον πάνω στη φυσική δημοκρατία σε αυτές τις χώρες. Πρόκειται οικονομικά προτεκτοράτα. Σε αυτό ε, μετατρέπονται αυτές οι χώρες ε, και διοικούνται από τον κύριο Μπαρόζο και τον κύριο Βαν Ρόμπαϊ. Τώρα έχουν δηλαδή μικρό αποτέλεσμα στις αποφάσεις τις οικονομικές τους. Είναι κάτω από τον έλεγχο των Βρυξελών, κάτω από τον έλεγχο των διεθνών οργανισμών. Όταν θα τελειώσει αυτή η κρίση πρέπει πραγματικά να αποκαταστήσουμε τη δημοκρατία σε αυτές τις χώρες ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να ελέγξουν την οικονομική τους πολιτική. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Μιγκουέλ Πόρτας, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην πολιτική πρέπει να πω ότι υπάρχουν λογικά μέτρα, λάθος μέτρα και δυσάρεστα μέτρα. Ε, είναι φυσικό να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό δημόσιο χρέος, έστω και αν η κυρία Μέρκελ δεν το θέλει. Είναι λογικό η Ευρώπη να θέλει να χρησιμοποιήσει, ε, ένα, ε, να καλύψει μάλλον ένα κομμάτι του δημοσίου αυτό που είναι δυσάρεστο όμως είναι να ακούμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τα Ευρωπαϊκά Ταμεία θα χρησιμοποιήσουν ένα τμήμα του, ε, ε, κρα, του κρατικού χρέους και θα το εξεγοράσουν από τις ιδιωτικές τράπεζες. Δηλαδή, έχουμε στην Πορτογαλία τράπεζες οι οποίες χρηματοδοτούνται από την ΕΚΤ με 1%. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι μέχρι πότε η Ευρώπη θα είναι ο δούλος του ε, διεθνούς κεφαλαίου. Μέχρι πότε θα μετατρέπουμε το, τα ιδιωτικά χρέη σε κρατικά, σε δημόσια. Μέχρι πότε οι φορολογούμενοι θα πληρώνουν τα χρέη των ιδιωτικών τραπεζών. Ο Μάριο Βοργέζιο τώρα για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, στη ΣΥΠΑ ένας νόμος επέβαλε στην ε, ΦΕΔ πόσα χρήματα θα δοθούν προς διάσωση ποιας τράπεζας. Ε, δεν θα μπορούσατε να έχετε τα ίδια κριτήρια διαφάνειας, εκτός αν το super lobby ε, το τραπεζικό σας το απαγορεύει έχουμε μία υποχρεωτική ένωση ελευθέρων χωρών. Ε, ε, οι ισχυρότερες χώρες έχουν στα χέρια τους τα χρέη των ασθενεστέρων. Το ευρώ είναι ένα νόμισμα που σχεδόν έχει πτωχεύσει. Πώς θα υποχρεώσουμε λοιπόν χώρες αδύναμες να το χρησιμοποιούν. Είναι αποδεκτή αυτή η πολιτική, η νομισματική, η κεντρική για χώρες που έχουν επιτόκια τόσο διαφορετικά. Ο ίδιος ο Τρισέ είπε ότι υπάρχει κίνδυνος αφαιρεγγιότητας της ΕΚΤ και πιστεύει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με μετακίνηση κεφαλαίων. Μιλάμε πάλι για στρες τεστ μεγάλων τραπεζών. Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο πρόεδρος, έχει λήξει ο χρόνος σας. Ο κύριος Κασουλίδης τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το μήνυμα από τις πολιτικό μήνυμα, Το πολιτικό μήνυμα από την τελευταία διάθεση κορυφής είναι ότι τα κράτη-μέλη θα κάνουν ό,τι χρειάζεται για να εξασφαλίσουν την Ευρωζώνη και να προασπίσουν το ευρώ. Όποιες και εσωτερικές συζητήσεις γίνονται κατά πόσον το δημοσιονομικό μέσο θα χρειαστεί να διπλασιάσει το κεφαλαίο του για να αγοράσει ομόλογα κατά πόσον μετά από το 2013 θα υπάρχει μείωση των ε, οικονομικών ή θα αγοραστούν τα ευρωομόλογα. Όλα αυτά δεν έχουν αποκλειστεί εκ των προτέρων από κανένα κράτος μέλος. Μόνο το χρονοδιάγραμμα συζητιέται. Τι χρειάζεται πότε. Οι αναλυτές δεν έχουν καμία, ε, κανένα πρόβλημα. Θα πάρει τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζεται η Ένωση όποτε χρειάζονται αυτά και όποια μέτρα. Όσον αφορά το μηχανισμό σταθερότητας, το Συμβούλιο λέει ότι θα πρέπει να κινητοποιηθεί ο μηχανισμό αυτό εάν είναι απολύτω απαραίτητο για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα του συνόλου τη Ευρωζώνη. Ως μέλος μιας, ε, από μια μικρή χώρα μέλος θα ήθελα να μου διαβεβαιώσετε ότι χώρες όπως η Μάλτα, η Εστονία, η Λετωνία και άλλες θα συμπεριληφθούν γιατί εάν εκείνες είναι, ε, έχουν πρόβλημα ίσως αυτό δεν είναι απαραίτητο για την σταθερότητα όλη της Ευρωζώνης. Η κυρία Πουδηματά ένα λεπτό οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι από την αρχή της κρίσης η ευρώπη αν και πλήρως απροετοίμαστη θεσμικά και πολιτικά έχει κάνει σοβαρά βήματα για να την αντιμετωπίσει από την εφαρμογή της δέσμης στήριξης της ελλάδας πριν από σχεδόν ένα χρόνο μέχρι τις αποφάσεις του τελευταίου ευρωπαϊκού συμβουλίου για τη σύσταση ενός μόνιμου μηχανισμού σταθερότητας έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς το εμπρός ωστόσο οι συνεχιζόμενες και διευρυνόμενες πιέσεις των αγορών και όχι πλέον μόνο σε βάρος των πλέον ευάλωτων οικονομιών της ευρωζώνης αποδεικνύουν ότι οι αποφάσεις μας είναι αποσπασματικές και είναι ανεπαρκείς για να δώσουν μια ολοκληρωμένη απάντηση στην κρίση. χρειαζόμαστε λοιπόν μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση που δεν θα υποκαθιστά ούτε θα παραβλέπει τις ευθύνες των κρατών μελών να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να εξηγειάνουν τα δημόσια οικονομικά τους αλλά θα προστατεύει τις οικονομίες αυτές από τις επιθέσεις των αγορών και θα διευκολύνει την ευόδοση των προσπαθειών τους. κύριε πρόεδρε το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με ψήφισμά του πριν από λίγες ημέρες ζητάει από την ευρωπαϊκή επιτροπή να προχωρήσει άμεσα σε μια μελέτη σκοπιμότητας για την έκδοση ευρωομολόγων. Η κυρία Φιγκερέδο έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Φτάσαμε στο τέλος της Ευρωπαϊκής Χρονιάς ε, αφιερωμένη στην καταπολέμηση της ένδυας ε, και του αποκλεισμού. Εάν κάνατε έναν απολογισμό θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν πάνω από 100 εκατομμύρια Φτωχή στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανεργία θα αυξήσει την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αλλά τα ε, και τα κέρδη των πολυεθνικών ε, και των κέρδοσκόπων αυξάνονται μέρα με την ημέρα βασιζόμενα στην πολιτικές της Κεντρικής Τράπεζας του Συμβουλίου και της Γι' αυτό έχουμε τη ζώνη ευρώ οι δράσεις κατά των πλέον αδυνάμων κρατών συνεχίζονται και οι κερδοσκόποι οργιάζουν. Θα πρέπει λοιπόν ε, να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται με τις εξελίξεις αυτές όπως συνέβη προσφάτω στην Πορτογαλία. Εμεί θέλουμε μια διαφορετική Ευρώπη, μια Ευρώπη τη κοινωνική προόδου που θα σέβεται του εργαζόμενου, και τα δικαιώματά τους. Μπορούμε να σας πούμε ότι εμείς θα είμαστε με την πλευρά των εργαζομένων. Το λόγο έχει ο κύριος Μίτσελ. Ε, oh, Δεν είναι εδώ ο κύριος Μίτσελ. Ο συνάδελφος Τιούν Κέλαμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που μπορώ να πω ότι είναι η 19η μέρα σήμερα της, από την ημέρα που έγινε η Εστονία μέλος του Ευρώ. Αλλά έχουμε προετοιμαστεί από τότε που προσχωρήσαμε. Συμφωνήθηκε ε, με τη λαϊκή ψήφο αυτό πριν από έξι χρόνια. Το να μπει κανεί όμως στην Ευρωζώνη δεν είναι προσωπική επιλογή, είναι επιλογή για περισσότερη αλληλεγγύη και για κοινή υπευθυνότητα ώστε να συμβάλλουμε σταθερά, ε, ε, συλλογικά στη σταθερότητα της Υπήρου στο σύνολό τη. Σε εποχή οικονομικής κρίσης οι ηθικές αξίες ενισχύονται. Το οικονομικό δυναμικό το ίδιο δεν αρκεί κρίσιμο είναι κατά πόσο θα έχουμε εμπιστοσύνη σε μια χώρα ότι θέλει να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της και στις υποχρεώσεις της εγκαίρως και ότι έχει πράγματι προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Χαίρομαι για το γεγονός ότι το Συμβούλιο συμφώνησε για το μηχανισμό σταθερότητας. Ένας πρακτικός τρόπος για οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα είναι να ολοκληρώσουμε πρώτα απ' όλα την ενιαία αγορά, ιδίως δε την ψηφιακή. Αυτή πρέπει να ενταχθεί στον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς καθώς και στην ψηφιακή ατζέντα. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματικά ευκαιρία προώθησης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στον κόσμο. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν να διευκολύνουμε την κατάσταση, την ψηφιακή, την ηλεκτρονική πληρωμή, την ταυτοποίηση. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν ομοιόμορφα και κατανοητά. Μία ενιαία ψηφιακή αγορά σημαίνει ανάπτυξη των υπεριών. Ευχαριστώ και τώρα ο Ζων Πιέρ μέσα στη διαδικασία Catch the Eye. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κύριε Μπαρόζο, κύριε Βαν ε, δύο σχόλια όσον αφορά την περίμετρο του μηχανισμού διαχείρισης της κρίσης. Για τα κράτη που δεν είναι μέλη της ζώνης έχουμε δύο κατηγορίες. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία που δεν είναι υποχρεωμένα να παίρνουν το ευρώ και τα άλλα κράτη που αποτελούν το σύνολο των 25. Θα ήθελα οι χώρες που είναι συνδεδεμένες με το ευρώ να έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση μέσα στο μηχανισμό. Επίσης θα ήθελα να επισύρω την προσοχή σας στα εθνικά κοινοβούλια. Στην απλουστευμένη διαδικασία δεν συμμετέχουν εκτός από την επικύρωση. Θα ήθελα να τα εντάξετε τα εθνικά κοινοβούλια στη διαβούλευση, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα ποιο θα κάνει τον πολιτικό έλεγχο του μελλοντικού μηχανισμού, το Ευρωκοινοβούλιο ή τα εθνικά κοινοβούλια. Και επειδή δεν έχουμε κοινοβουλευτική διάσταση της Ευρωζώνης, δεν ξέρουμε πώς θα ελέγξουμε πολιτικά αυτό τον μηχανισμό. Σας υποβάλλω τι σκέψει μου. Ευχαριστώ ο Ρομπέρτι Γκάου Γκαλτιέρη. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε του Συμβουλίου. Εγώ διακρίνω δύο μεγάλα προβλήματα σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 136, ένα θεσμικό και ένα πολιτικό. Το θεσμικό, το άρθρο 3 τη συνθήκη σχετικά με τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση προσδιορίζει την ε, νομισματική πολιτική του, Ένωση για το ευρώ, που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα. Αλλά το άρθρο παρακάτω αναφέρει ότι μπορεί να ε, γίνει, εφαρμοστεί αυτή η πολιτική αν ε, δοθεί άδεια από τα κράτη-μέλη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας κανόνας που περιλαμβάνεται στις συνθήκες απαιτεί ταυτόχρονα και μια μεταρρύθμιση. Αυτό είναι ένα πολιτικό πρόβλημα. Το πολιτικό πρόβλημα ποιο είναι, η επιλογή της ε, τροποποίησης συνθήκης, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 2 ή το 322, θέτει το μέλλον του ευρώ στο πλαίσιο της διαδικασίας επικύρωσης από 27 κράτη-μέλη. Εάν λοιπόν μία από αυτές τις διαδικασίες επικύρωσης δεν προχωρήσει θα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί ένα σχέδιο ε, για ε, ε, αναπληρωματικό προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Γκαλπέτζου. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Η σταθερότητα του ευρώ και η ε, επίλυση της κρίσης ε, είναι ένα από τα άμεσα καθήκοντά μας. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης και να περιορίσουμε το χρέος των κρατών. Όλοι φυσικά συμφωνούμε πάνω σε αυτό, αλλά προσπαθώντας να ξέρουμε λύση, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα, κάποια στρατηγικά ζητήματα όπως αυτό της καινοτομία. Είχαμε ήδη μια συζήτηση τον Δεκέμβριο. Η επόμενη σύνοδος του Συμβουλίου τον Φεβρουάριο θα πρέπει να λάβει σημαντικές αποφάσεις όπως στο ζήτημα της ενέργειας. Η Ουγγρική Προεδρία ξεκίνησε ήδη αυτή την διαδικασία. Οι βασικότεροι κανόνες υιοθετήθηκαν πέρυσι, όπως ο κανόνας σχετικά με την προμήθεια σε φυσικό αέριο και τον εφοδιασμό της Ένωσης, Πρόεδρε. Ελπίζω αυτά τα ενεργειακά προβλήματα να μην παραμεριστούν λόγω των άλλων ζητημάτων. Ως γνωστόν για δεύτερη φορά στην παρούσα χρηματοπιστωτική κρίση η κυβέρνηση των ηνωμένων πολιτειών αναγκάστηκε εξ αρχής σε δραματική παρέμβαση για να στηρίξει τις δύο μεγάλες τράπεζες που κατέρεαν και τον ασφαλιστικό οργανισμό ang. έτσι προσέφερε 700 δις οικονομική βοήθεια στο παράλληλο το τραπεζικό της σύστημα. παρά τα μέτρα αυτά η οικονομία των ηπα χρειάστηκε και άλλη βοήθεια και χωρίς φιδό η κυβέρνηση προσέφερε πρόσφατα επιπλέον κεφάλαιο 600 δις δολαρίων προκειμένου η οικονομία να βγει από την ύφεση. είναι σαφέ ότι οι ηνωμένε πολιτείε εκδίδουν νέο χρήμα κύριε πρόεδρε. σε αντίθεση με την οικονομία των ηπα η ευρωζώνη παραμένει σταθερή στην αρχή τη δημοσιονομική πειθαρχία, στην αυστηρώ ελεγχόμενη νομισματική πολιτική με αποτέλεσμα να αφήνει χώρο στι ε, κερδοσκοπικές διάφορες επιχειρήσεις να κερδοσκοπούν σε βάρο των λιγότερο ανθεκτικών στι πιέσει κρατών κύριε πρόεδρε προτείνω να εξετάσουμε την έκδοση νέου χρήματος στην ευρωζώνη. ίσως είναι το αυγό του κολόμβου. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Η κυρία Λίζα Γιακονσάρη. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει σπάθα του ε, δαμόκλειο σπάθα πάνω από την Ευρώπη. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα φύγουμε. Η ομάδα μου αναρωτιέται κατά πόσον η Ευρώπη μπορεί να ενωθεί όταν υπάρχει ε, μια βοήθεια από τις ιδρυτικές χώρες ή υπάρχει αυτό το ε, αυτός ο κίνδυνος της ε, διάσπασης και του καταγερματισμού. Αναρωτιέμαι, είναι περίεργο ότι είμαστε τόσο αδύναμοι εδώ, γιατί δεν τίθεται το θέμα κατά πόσον η πολιτική ε, οδηγεί τις αγορές ή οι αγορές οδηγούν την πολιτική. Η πολιτική είναι στο δρόμο, η πολιτική είναι σε διαδηλώσεις από ακραίες ομάδες του πληθυσμού. Και γι' αυτό θα πρέπει τα κοινωνικά θέματα να είναι αυτή τη στιγμή τα πιο σημαντικά για την Επιτροπή, αλλά δυστυχώ δεν γίνεται τίποτα στο τομέα αυτό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ο κύριο Σον Κέλλη έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω και άλλοι, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Φανερόπα και τον κύριο Παρόζο που τουλάχιστον προσπαθούν να δράσουν στη σημερινή κρίση και εισαγάγουν μέτρα που ελπίζουμε ότι θα είναι επιτυχή στο μέλλον. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή βέβαια να πούμε κατά πόσο θα είναι αυτό ε, πραγματικό. Εάν ε, επιτύχουν θα είναι ήρωες, εάν όχι θα είναι οι κακοί. Θα πρέπει να έχουμε μια σοφή δομή, ούτως ώστε ε, τα περισσότερα σφάλματα που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση θα υπάρχουν και στο μέλλον. Όσον αφορά τις ανησυχίε της δικής μας χώρας, υπήρχαν κάποιες προσπάθειες διάδοσης για μια κρίση στην οποία οδήγησαν προβλήματα των τραπεζών. Εγώ θα ήθελα να κάνω έκκληση στους κυρίους Φερνόπα και Μπαρόσο να μειώσουν τα επιτόκια που ζητούνται για τα δάνεια αυτά γιατί είναι πολύ ψηλά και καταστρέφουν τις οικονομίες περαιτέρω. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα αυτή η συζήτηση κατέδειξε πόσο περίπλοκο, περίπλοκη είναι η κρίση και πόσο περίπλοκες είναι και οι απαντήσεις. Ένα πράγμα που θα ήθελα να πω σε εκείνους και είναι σαφώς η μεγάλη πλειοψηφία που συμμερίζονται τα ευρωπαϊκά ιδανικά και θέλουν μια ευρωπαϊκή απόκριση είναι ότι δεν πρέπει να χωριζόμαστε με κάποιες διαφορές οι οποίες δεν είναι σημαίνουσες. Όπως είπατε ορισμένοι, υπάρχει μια πραγματική πρόκληση και μάλιστα και θα έλεγα και απειλή για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Την έχουμε δει αυτή την απειλή στη συζήτηση αυτή. Άκουσα κάποια σχόλια νασιοναλιστικά, εθνικιστικά, που ειλικρινά δεν τα έχω συνηθίσει να τα ακούω σε αυτό το κοινοβούλιο. Είναι μειοψηφία βέβαια ε, από μειοψηφία έγιναν αυτά τα, σχόλια, τα οποία όμως θέλουν να εμβαθύνουν τις διαφορές μεταξύ των λεγόμενων πλουσίων και φτωχών Ευρωπαίων. Σε όσο έκαναν αυτά τα σχόλια κατά της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, προσπαθώντας να εμβαθύνουν το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, θέλω να τους ρωτήσω αυτούς Πού ήσασταν όταν χρηματοδοτούσε η Ευρώπη τους αγρότες σας για να ταΐσει τον λαό σας. Πού ήσασταν όταν η Ευρώπη χρηματοδοτούσε τις υποδομές σας για να αναπτυχθεί και να γίνει ανταγωνιστική η χώρα σας. Πού ήσασταν όταν η Ευρώπη δημιούργησε την εσωτερική αγορά για να πουλάτε τις υπηρεσίες σας και τα προϊόντα σας. Πού ήσασταν όταν η Ευρώπη ήταν η βάση για την ευημερία και την ανάπτυξη των χωρών σας μετά τον πόλεμο. Μόνο εγωιστές, κοντόφθαλμοι στις απόψεις τους μπορούν να έχουν, κάνουν τέτοιες δηλώσεις κατά της Ευρωπαϊκής Ενότητας και νομίζω είναι, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, το θίξατε πολύ από εσά. Κάνω έκκληση λοιπόν σε όσους συμμερίζονται τα ευρωπαϊκά ιδανικά. Ενωθείτε. Δημιουργήστε μία συντονισμένη απόκριση σε ένα θέμα που είναι σοβαρό. Πρέπει να δημιουργηθεί συνένεση και καμιά φορά ομολογουμένως δεν είναι εύκολη η συνένεση σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με 27 χώρες, μια Ευρωζώνη με 17 χώρες και καλωσορίζω την Εστονία, το νέο μέλος και μια διαδικασία λήψης απόφασης που δεν είναι πάντοτε η πιο απλή διότι βασίζεται στις αρχές της δημοκρατίας και ε, έχουμε 27 δημοκρατίες και όλους τους θεσμούς ευρωπαϊκούς. Είναι πολύ δύσκολο το έργο, αναμφίβολα. Γι' αυτό κάνω έκκληση προς όλους όσους συμμερίζονται τα ευρωπαϊκά ιδανικά. Μην χάνουμε το δρόμο μας με κάποιες μικροδιαφορές. Κύριε Στέφεν Ιούς, ε, ε, αντιλαμβάνομαι πλήρως την κοινωνική χρειά της Ευρώπης, αλλά να είμαστε σαφείς. Πώς μπορούμε καλύτερα να υποστηρίξουμε κυβερνήσεις όπως την ελληνική κυβέρνηση, την ισπανική κυβέρνηση, την πορτογαλική κυβέρνηση που έχουν πολύ σημαντικούς πολιτικούς ηγέτες να υποστηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις τους τις τολμηρές ή να πούμε απλά ότι αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι κατά των ευρωπαϊκών αξιών. Χρειαζόμαστε ε, διαρθρωτικ κατά μία και στον τομέα της απασχόλησης στην Ευρώπη. Αν ρωτήσετε τον Πρωθυπουργό Παπανδρέου, Σόκρατε, Ζαπατέρο, ακριβώς αυτό κάνουν και έχουν σκοπό να πάνε ακόμη βαθύτερα στις μεταρρυθμίσεις. Λοιπόν, πραγματικά πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος να υποστηρίξουμε τις θαραλές προσπάθειες της Ευρώπης είναι να χρησιμοποιούμε τη γλώσσα της αλήθειας στον σημερινό κόσμο του ανταγωνισμού με την πίεση των αναδειωμένων οικονομιών που γίνονται ισχυρότερες θα διακινδυνέψουμε την κοινωνική οικονομία αγοράς που έχουμε. Δεν αμφισβητούμε τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Θα απαντήσω εδώ και σε εσά ένα λεπτό. Δεν σας έχω ξεχάσει την ερώτησή σας. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να σεβόμαστε τα, τις αρχές του κοινωνικού διαλόγου. Το είπα χθε, το ξαναλέω και σήμερα. Όμως, εάν δεν κάνουμε την φορολογική παγίωση και την δημοσιονομική μεταρρύθμιση, δεν θα έχουμε εμπιστοσύνη και χωρίς το εμπιστοσύνη δεν θα έχουμε ανάπτυξη και συνεπώς δεν θα έχουμε απασχόληση για τους πολίτες μας. Λοιπόν, όσον αφορά τον εκλεκτό βουλευτή από την Ιρλανδία, που είπε ότι τα προβλήματα της Ιρλανδίας θα δημιούργησε η Ευρώπη θα σας πω ότι ήταν ανεύθυνη η συμπεριφορά ορισμένων Ιρλανδικών οργανισμών. Η Ευρώπη και από εκεί δημιουργήθηκε το πρόβλημα της Ιρλανδίας. Και σήμερα η Ευρώπη είναι κομμάτι της λύσης. Υποστηρίζει την Ιρλανδία και δεν είναι η Ευρώπη που δημιούργησε αυτή την απαράδεικτη φορολογική κατάσταση. Η Ευρώπη προσπαθεί να υποστηρίξει την Ιρλανδία. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε πού βρίσκεται η ευθύνη. Και γι' αυτό είναι εξίσου σημαντικό όσοι από εμά και έχουμε την πλειοψηφία πιστεύουμε στα ευρωπαϊκά ιδανικά να μπορέσουμε να οργανώσουμε μια κοινή απόκριση. Ένα άλλο σχόλιο που κάνατε είναι ε, ποιο είναι το επίπεδο της φιλοδοξίας. Θα είμαι σαφής για την Κομισιόν. Είμαστε για την πιο φιλόδοξη θέση όσον αφορά μια ολοκληρωμένη απόκριση. Γι' αυτό η Κομισιόν θα είναι έτοιμη να υποστηρίξει μέτρα που ορισμένοι από εσά έχετε προτείνει. Όμως έχουμε την εξής κατάσταση. Σε περίπτωση κρίσης σαν και αυτή και σε αστάθεια των αγορών είναι πολύ σημαντικό να συμβάλλουμε σε συνένεση όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Υπήρξαν διαφορές όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης αυτής της κρίσης μεταξύ κρατών μελών. Αναθεώρηση τώρα της συνθήκης. Ξέρετε ποια ήταν η θέση της Κομισιόν. Είπαμε εξ αρχής ότι πιστεύαμε ότι ήταν δυνατόν να δημιουργήσουμε ένα μόνιμο μηχανισμό χωρίς τροποποίηση. Όμως ένα κράτος μέλων, μέλος σαφώς είπε και χρειαζόμαστε ομοφωνία σαφώς είπε ότι θέλει τροποποίηση και εφόσον είναι σημαντικό να έχουμε ένα μόνιμο μηχανισμό η Κομισιόν ήταν επικοδομητική και υποστήριξε αυτή την περιορισμένη τροποποίηση. Θα ήταν τελείως λάθος λοιπόν να έχουμε διαφορετικές θέσεις σε αυτό το θέμα. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη σταθερότητα. Είναι συνεπώς σημαντικό να συμφωνήσουμε για αυτή την περιορισμένη αναθεώρηση της συνθήκης. Ορισμένοι θα θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο. Και εγώ θα προσωπικά θα το ήθελα όσον αφορά την αναδιάρθρωση της κοινοτικής προσέγγισης. Θα πρέπει όμως να είμαστε υπεύθυνοι σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που ζούμε πρέπει να βρούμε τον υψηλότερο κοινό παρανομαστή, όχι τον χαμηλότερο. Και γι' αυτό δηλώνω και πάλι ότι ορισμένε από τις προτάσεις που έγιναν ε, είναι καλές οι ίδιες, αλλά δεν μπορούν να ε, προκαλέσουν σήμερα συνένεση. Και γι' αυτό πρέπει η Κομισιόν να ασχολείται με τη σφυριλάτηση της συνένεσης δεν μ' αρέσουν καθόλου οι διαχωρισμοί μεταξύ πλουσίων και φτωχών, κέντρου και περιφέρειας. Ε, στην Ευρώπη όλα τα κράτη έχουν ακριβώς την ίδια αξιοπρέπεια. Οι ιδέες ε, εφαρμογής διακρίσεων μεταξύ των κρατών μελών είναι πολύ επικίνδυνες για το ευρωπαϊκό σχέδιο. Πώς λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε θα πρέπει να ρωτήσουμε όλα τα κράτη-μέλη που είναι σε ευάλωτη κατάσταση να πράξουν ό,τι χρειάζεται για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην οικονομία τους μέσω του μηχανισμού σταθερότητας, της αναδιάρθρωσης των δομών, της φορολογικής μεταρρύθμισης. Δεν βοηθάμε αυτές τις χώρες αν τους λέμε ότι μπορεί να διαφύγουν. Ταυτόχρονα αυτές οι χώρες που είναι σε καλύτερη κατάσταση πρέπει να επιδείξουν αλληλεγγύη προς τους ευάλωτους. Είναι σημαντικό να έχουμε σημαντική απόκριση όσον αφορά τη σταθερότητα του ευρώ. Ε, όχι μετά τη στροφή, αλλά πριν από τη στροφή. Δηλαδή να έχουμε μία ε, συντονισμένη απόκραση από τις χώρες του ευρώ και από την Ένωση μέσω πράξεων, όχι μόνο μέσω δηλώσεων. Οι δηλώσεις είναι σημαντικές αλλά δεν είναι απαρκείς, είναι σημαντικές οι ενέργειες και σαν σύνολο όλοι μας. Πρέπει να δεσμευτούμε για ισχυρότερη διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη και στην Ένωση. Αυτό μας ζητούν οι αγορές. Υπάρχει πρόβλημα με το πώς γινόμαστε αντιληπτοί. Δηλαδή πώς μπορούμε να λάβουμε αποφάσεις και να τις αφαρμόσουμε. Χρειαζόμαστε ενισχυμένη διακυβέρνηση με καλύτερο συντονισμό και βασικά όλοι μας πρέπει να δεσμευτούμε για αλληλεγγύη και υπευθυνότητα. Δεν είναι μόνο θέμα υπευθυνότητας. Υπάρχει και το θέμα της αλληλεγγύης. Δεν είναι μόνο θέμα αλληλεγγύης, υπάρχει και θέμα υπευθυνότητας. Λοιπόν, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε σταθερότητα και η σταθερότητα είναι η βάση για τη μελλοντική μας ευμερία. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο πρόεδρος Σέλμαν Φανρόπο έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάλφοι, θα ξεκινήσω με κάποια θετικά στοιχεία. Καταρχήν η οικονομική ανάκαμψη είναι πολύ ισχυρότερη από ό,τι πιστεύαμε πριν από μερικές εβδομάδες ή μήνες. Πολύ πιο ισχυρή. Σε ορισμένα κράτη η ανεργία μειώνεται. Ποιος θα πίστευε κάτι τέτοιο το 2008 και το 2009. Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2010-2011 η απασχόληση θα αυξηθεί εκ νέου μετά από την σημαντικότερη κρίση τα τελευταία 70 έτη. Πάνω σε αυτό σίγουρα κανείς ε, δεν θα είχε συμφωνήσει αλλά η πραγματικότητα αυτή είναι φυσικά υπάρχει κρίση αλλά το κοινό νόμισμα των 17 κρατών μιλών παραμένει σταθερό σε σχέση με το ευρωπαϊκό δολάριο και η ισοτιμία είναι 1,30 στο παρελθόν είχε φτάσει το 0,80 ουδής τότε είχε δηλώσει πως το ευρώ κινδύνευε σε σχέση με άλλες επίρους και άλλα μεγάλα νομίσματα έχουμε ένα ισοζύγιο πληρωμών στις τρέχουσες συναλλαγές που βρίσκεται σε ε, που είναι ίσως και σε σχέση με άλλα κράτη έχουμε ένα έλλειμμα το οποίο έχει μειωθεί. Αυτό εξηγεί ότι παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, το Ευρώπη είναι ένα νόμισμα σταθερό. Θα ήθελα να τονίσω αυτά τα στοιχεία προτού να περάσω στα υπόλοιπα. Φυσικά και γνωρίζουμε πως πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά χρειάζεται να θυμηθούμε, όπως είχα πει εξάλλου και στην τελευταία μας συνάντηση εδώ στο Κοινοβούλιο, αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκίνησε αυτή η κρίση της Ευρωζώνης που είναι περισσότερο κρίτη της Ευρωζώνης και όχι του ευρώ, δίχως ε, κατάλληλα μέσα, κατάλληλα εργαλεία. Χρειάστηκε να εφεύρουμε κάποια εργαλεία. Αυτό εξηγεί και τον λόγο για τον οποίο δεν προχωρήσαμε αρκετά γρήγορα από ό,τι επιθυμούσαμε και από ό,τι απαιτούσαν οι συνθήκες και η συγκυρία αλλά δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη, το οποίο όμως δεν ετηρείτο. Δεν υπήρχε μακροοικονομική εποπτεία, δεν είχαμε μηχανισμό κρίσης ούτε προσωρινό ούτε σταθερό και δεν υπήρχαν ισχυρά θεσμικά όργανα για την δημοσιονομική εποπτεία. Χρειάστηκε όλα να τα εφεύρουμε καθοδόν. Και αυτό είναι ένα ζήτημα συλλογική ευθύνη Ορισμένοι ημών είπαν ότι είναι πολύ λίγα και φτάνουν πολύ αργά. Too little and too late. Αλλά το γεγονός ότι δεν είχαμε κανένα εργαλείο εξηγεί το ότι δεν βρισκόμαστε στο too little too late αλλά στον, στην ε, φάση βήμα προς βήμα. Ορισμένοι εξημών επίσης είπαν ναι, μα η κρίση δεν βρίσκεται υπό έλεγχο. Κοιτάξτε τι γίνεται με τις ε, αγορές. Αλλά ταυτόχρονα άλλοι, αλλά και συχνά οι ίδιοι δηλώνουν ότι δεν μπορούν οι αγορές να υπαγορεύουν τη δράση σας. Είτε το ένα θα ισχύει είτε το άλλο. Αλλά δεν υπάρχει πάντα συνέπεια μεταξύ αυτών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα τα οποία λάβαμε, φυσικά ε, υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που πρέπει να ξεκινήσουν στα κράτη-μέλη, όχι μόνο στις χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά σε όλα τα κράτη-μέλη. Μεταρρυθμίσεις για να απελευθερώσουμε το δυναμικό της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Και φυσικά οι μεταρρυθμίσεις ψηλά είναι, είναι επίπονες Χρειάζεται λοιπόν να εργαστούμε σωστά για να υπάρξει μια δίκαιη κατανομή των προσπαθειών που απαιτούνται. Να υπενθυμίσω ότι η, μια μεγάλη χώρα εξέρχεται πιο γρήγορα από την οικονομική κρίση και έλαβαν μέτρα όμως πριν από 5 ή 6 χρόνια αυστηρά και τότε υπήρξαν σημαντικές αντιδράσεις από το σύνολο του κοινωνικού ιστού. Αλλά αυτό δημιούργησε επιπτώσεις και συνέπειες τόσο σε ό,τι φορά την ανάπτυξη όσο και την απασχόληση. Χρειάζεται λοιπόν να φτάσουμε σε κρίσιμο σημείο, στον πάτο θα λέγαμε του βαρελιού, για να μπορέσουμε μετά να ανεβούμε τον δρόμο και να επανέλθουμε στην ε, οδό της ανάκαμψης και της ανάπτυξης. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις λοιπόν σε ε, επίπεδο κρατών μελών, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης ιδιαίτερα. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία να εφαρμόσουμε το συντομότερο δυνατόν την οικονομική διακυβέρνηση που αποφασίσαμε στην Task Force και που συζητήσαμε με βάση τις έξι προτάσεις της Κομισιόν εδώ στο Κοινοβούλιο και να εξεύρουμε λύση μεταξύ των εμπλεκομένων στο πλαίσιο της συναπόφασης. Είναι κάτι το ιδιαίτερα επίγον. Εάν είναι απαραίτητο να πάμε ακόμα παραπέρα, στο πλαίσιο της Ευρωζώνης σε ό,τι φορά τη σύγκληση της οικονομικής ανάπτυξης και των οικονομικών πολιτικών πρέπει να το πράξουμε. Εάν μπορούμε να το πράξουμε μέσω συμφωνιών ανάμεσα στα κράτη-μέλη στην Ευρωζώνη, θα πρέπει όχι μόνο να το σκεφτούμε, αλλά θα πρέπει να δουλέψουμε προκειμένου να ολοκληρώσουμε το έργο μας μέσα σε μερικές εβδομάδες ή και μήνες. Αλλά ίσως να χρειαστεί να πάμε ακόμα παραπέρα στο πλαίσιο της Ευρωζώνης από αυτά που αποφασίστηκαν στην Task Force και που περιέχονται στις προτάσεις της Κομισιόν διότι ε, όταν έχουμε ένα κοινό νόμισμα χρειαζόμαστε και κοινέ οικονομικές πολιτικές και οικονομικές ε, και οικονομικής ανάπτυξης ε, κοινέ σε όλες τις χώρες της Eurozone. Ξεχάσαμε την διαθροντική οικονομική ανάπτυξη, όχι. Γι' αυτό και αποφασίσαμε για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2020. Περί αυτού θα συζητήσουμε σε μερικές εβδομάδες το Συμβούλιο του Φεβρουαρίου σχετικά με την καινοτομία και την ενέργεια, διότι μεταξύ όλων των προβλημάτων δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις ε, προοπτικές, τις πιο μακροπρόθεσμες, ε, τις διαφορετικές ε, πολιτικές ανάπτυξης και απασχόλησης. Και, σε, και βράχει πρόθεσμα προετοιμάζουμε μια σφαιρική προσέγγιση για την ενίσχυση των μέσων που δημιουργήσαμε το 2010 για να ξεπεράσουμε την κρίση και να την αντιμετωπίσουμε. Έχουμε μια ατζέντα σαφή. Μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα, να αυξήσουμε ταχύτητα, ναι. Αλλά σας είπα υπάρχουν δύο προβλήματα, υπήρχαν δύο προβλήματα. Πρώτον, ότι χρειάστηκε να τα ε, βρούμε όλα και να τα φτιάξουμε καθοδόν διότι και μια που βρισκόμαστε στη δημοκρατία χρειάζεται και απαιτείται ε, συνένεση από τα 27 κράτη-μέλη. Αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι υποστηρίζουν το ευρωπαϊκό σχέδιο αποτελούν την πλειοψηφία σε αυτό το κοινοβούλιο. Ας μην ε, ε, κάνουμε συναγωνισμό ποιος είναι ο πιο ευρωπαϊστής Νομίζω ότι έτσι θα δημιουργήσουμε μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα στους ε, υποστηριχτές και τους, ε, τους διασώτες και τους αντιπάλους Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε την κατεύθυνση, την πορεία, τον προσανατολισμό. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από ότι τα επιμέρους βήματα. Είναι η κοινή βούληση του να εργαστούμε προς την αυτή κατεύθυνση για την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού σχεδίου που είναι θεμελιώδους και κεφαλαίωδους σημασίας που επαναλήφθηκε και στην ε, Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Γι' αυτό λοιπόν με αυτή την προσέγγιση βήμα προς βήμα θα το πετύχουμε. Είμαι πεπισμένος ότι βρισκόμαστε στην σωστή πορεία, είμαι πεπισμένος ότι υπάρχει κοινή βούληση και είμαι πεπισμένος ότι επιτέλους θα το πετύχουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε για την παρουσίαση αυτή. Η επόμενη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα είναι στις 4 Φεβρουαρίου και κατόπιν αυτού βέβαια πάλι το Φεβρουάριο η επόμενη παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τον Πρόεδρο Φανρόποη. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και πρωτού περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης που είναι η ε, Ουγγρική Προεδρία. Δύο λεπτά διακοπή, μόνο δύο λεπτά.